Αγαπητοί συνάδελφοι, τώρα θα ψηφίσουμε για την εκλογή των κοσμητόρων. Έχουμε πέντε θέσεις με εφτά υποψηφίους. Και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. οι ψηφολέκτε θα είναι, η φορευτική επιτροπή θα είναι ίδια με τους ε, χθεσινούς. Είναι εδώ η συνάδελφος Μπορσελίνο. Σόγκορ. Παναγιώτοφ. Δεν είναι. αντικαταστάθηκε από την κυρία Πακ μου λένε. Ε, κυρία Πακ, κύριε Πρόεδρε, σήμερα το πρωί μόνο ε, αντικατέστησα τον συνάδελφο, γιατί σήμερα, ξέρετε, τώρα έχω και μια ομάδα επισκεπτών. Παρακαλώ κάποιον άλλο συνάδελφο να αναλάβει. Μα λύθηκε, λύθηκε το πρόβλημα, διότι ο κύριος Παναγιώτος εδώ είναι. Οπότε μπορεί να κάνει τη δουλειά του. Ποκ, μπαγκό. Παρόν. Καλινόφσκι. Ωραιότατα. Κάλφιν. Περέιρο Ροντρίγες. Ή η κυρία Μπορσελίνο. Εδώ είναι. Ωραία. Άρα έχουμε την εφορευτική. Παρακαλώ, ελάτε ο καθένας στα, κοντά στις κάλπες, μοιράστε τα ψηφοδέλτια, αν δεν έχουν μοιραστεί. Παρακαλώ. Μοιράστε τα ψηφοδέλτια. Από τώρα μπορούμε να ψηφίσουμε. Ξεκινάει η ψηφοφορία τώρα.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 Cinque voti. Πέντε, πέντε. Πέντε μπορείτε να ψηφίσετε. Ονορεύολε Σιλβέστρη. Κύριε Σιλβέστρης, πέντε μπορείτε, μπορείτε να ψηφίσετε.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 Ευχαριστώ. Μπορούμε να θεωρήσουμε λήξασα την διαδικασία ψηφοφορίας για τους κοσμήτορες θα συνεχιστεί η Ολομέλεια στις 3.